Dear <clears throat> Αγαπητοί συνάδελφοι, πάμε στο πρόγραμμά μας. Έχουμε τρεις εκθέσεις να ψηφίσουμε. Να είστε έτοιμοι λοιπόν με τις κάρτες σχέδιο γνωμοδοτήσεως για την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων στα πλαίσια της συνθήκης της Λισαβόνας από τον εισηγητή τον κύριο Άντριο Νταφ. Το συζητήσαν το θέμα το πρωί. Και πάμε στην ψηφοφορία τροπολογία 1 υπέρ Απερίφθη. 2 υπέρ. Απορρίπτεται. 3 υπέρ. Εγκρίνεται. 4 υπέρ. Εγκρίνεται. 5 υπέρ. Εγκρίνεται. 6 υπέρ. Εγκρίνεται. 7 υπέρ. Ε, απορρίπτεται. 8 υπέρ. Εγκρίνεται. 9 υπέρ. Εγκρίνεται. 10 υπέρ. 9. Την 9 να ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 9. Ξεκινάμε την ψηφοφορία. 9. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος ψηφοφορίας. Και το αποτέλεσμα είναι απόρριψης. 10 υπέρ. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία που αφορά την παράγραφο 12. Υπέρ εγκρίνεται. Πάμε στη 12. Συγγνώμη, αποσύρεται 13 υπέρ. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος, μάλλον ψηφίζουμε την γνωμοδότηση που ξεκινάει, ηλεκτρονική ψηφοφορία, τέλος και το αποτέλεσμα είναι 33 ψήφοι υπέρ, 4 ψήφοι κατά. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον κύριο Άνδριο Νταφ. Ελέγχω, όχι. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στο σχέδιο γνωμοδοτήσεως για τις δημοσιονομικές πτυχές της μεταρρυθμιστικής συνθήκης του Ιστβαν Σεντιβάνη και πρέπει να ψηφίσουμε τρεις τροπολογίες. Την ένα υπέρ απορρίπτεται. Δύο υπέρ απορρίπτεται. Τρία υπέρ απορρίπτεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία του σχεδίου γνωμοδοτήσεως τροποποιήθη. Ξεκινάμε. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Και το αποτέλεσμα είναι 32 ψήφι υπέρ, 6 κατά και συγχαρητήρια στον κύριο Σαντιβάνη. Εγκρίθηκε. Πάμε σε περιπλοκότερη ψηφοφορία. Σχέδιο εκθέσεως για την κατάσταση των διατλαντικών ε, σχέσεων μετά τις αμερικανικές εκλογές του κυρίου Φρανσίσκο Χωζέ Μιλανμόν. Χωζέ. Χωσέτ Χωσέ. Τα ανακατεύω τα πορτογαλικά μου, βλέπετε με μπερδεύουν. Ζωζή στα πορτογαλικά. Ζωζή Ντουράου. Καλώ. Ψηφίζουμε τώρα. Τροπολογία 42 υπέρ. Εγκρινάται. Συμβιβαστική 1 υπέρ. Εγκρινάται. Συμβαστική 2 υπέρ. Εγκρίνεται. 48 υπέρ. Απορρίπτεται. 49 υπέρ. Απορρίπτεται. 53 υπέρ. Απορρίπτεται. 54 υπέρ. Απορρίπτεται. 55 υπέρ. Απορρίπτεται. 56 και 57 υπέρ απορρίπτονται 58 ναι 58 υπέρ απορρίπτεται 59 υπέρ απορρίπτεται 60 υπέρ απορρίπτεται 61 υπέρ εγκρίνεται 62 υπέρ απορρίπτεται 63 υπέρ απορρίπτεται 64 υπέρ. Απορρίπτεται. 65 υπέρ. Απορρίπτεται. 66 δεν ψηφίζουμε. 67 υπέρ. Εγκρίνεται. 68. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Εγκρίνεται. με προφορική τροπολογία όσο αναφέρεται. Μάλιστα. Πάμε στην 73 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα της 73 υπέρ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Απορρίπτεται. Πάμε στη συμβαστική 4 με προφορική υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Εγκρίνεται. 51 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Εγκρίνεται. 82 σε δύο τμήματα, αλλά δεν ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα, ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα υπέρ. Εγκρίνεται. 83 υπέρ. Απορρίπτεται. 84 υπέρ. Απορρίπτεται. 85 υπέρ. Απορρίπτεται. 86 υπέρ. Εγκρίνεται. 87 υπέρ, εγκρίνεται. 88 υπέρ, εγκρίνεται. 89 υπέρ, απορρίπτεται. 90 υπέρ, εγκρίνεται. 91 υπέρ, απορρίπτεται. 92 υπέρ, απορρίπτεται. 93 υπέρ, απορρίπτεται. 94 υπέρ, απορρίπτεται. 95 υπέρ, εγκρίνεται. 96 υπέρ, απορρίπτεται. 97 υπέρ, εγκρίνεται. 98 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Εγκρίνεται. 99 υπέρ. Απορρίπτεται. 100 υπέρ. Κατά. Να γίνει έλεγχος για την 100. Παρακαλώ ψηφίστε. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Το αποτέλεσμα είναι 21 ψήφοι υπέρ, 23 κατά, απορρίπτεται κατά δύο ψήφους. Συμβαστική 6 υπέρ. 110 υπέρ. Εγκρίνεται. 111 υπέρ. Απορρίπτεται. 112 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ απορρίπτεται 113 13-14 Δεν ψηφίζουμε την 113 114 υπέρ απορρίπτεται 115 με προφορική υπέρ εγκρίνεται 116 υπέρ εγκρίνεται. 117 υπέρ, απορρίπτεται. 118 υπέρ, καλύπτεται. 119 υπέρ, απορρίπτεται. 120 υπέρ, απορρίπτεται. 121 υπέρ, εγκρίνεται. 122 υπέρ, απορρίπτεται. 123 υπέρ, απορρίπτεται. 124 υπέρ, εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ εγκρίνεται. 134 υπέρ απορρίπτεται. 135 υπέρ κατά. Έλεγχος για την 135 ηλεκτρονική ψηφοφορία που ξεκινάει. 135 ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Το αποτέλεσμα είναι 24 με 19 εγκρίνεται και πάμε στην 136 υπέρ εγκρίνεται 137 υπέρ απορρίπτεται 138 υπέρ απορρίπτεται 139 υπέρ απορρίπτεται 140 υπέρ απορρίπτεται 141 υπέρ απορρίπτεται 142 υπέρ απορρίπτεται 143 υπέρ εγκρίνεται 144 υπέρ απορρίπτεται 145 υπέρ απορρίπτεται 146 υπέρ απορρίπτεται 147 υπέρ απορρίπτεται 148 υπέρ καλύπτεται συγγνώμη 149 υπέρ απορρίπτεται 150 υπέρ απορρίπτεται συμβαστική 9 υπέρ εγκρίνεται 156 υπέρ απορρίπτεται 157 υπέρ απορρίπτεται 158 υπέρ απορρίπτεται 159 υπέρ απορρίπτεται 160 υπέρ εγκρίνεται 161 υπέρ εγκρίνεται 162 υπέρ εγκρίνεται 163 υπέρ εγκρίνεται 164 υπέρ απορρίπτεται 165 υπέρ εγκρίνεται προφορική τροπολογία που αφορά την παράγραφο 35 υπέρ εγκρίνεται 166 υπέρ εγκρίνεται 167 υπέρ εγκρίνεται 168 υπέρ εγκρίνεται 169 υπέρ εγκρίνεται αιτιολογική σκέψη α τροπολογία 4 υπέρ Απορρίπτεται. 5 υπέρ. Απορρίπτεται. 6 υπέρ. Απορρίπτεται. 7 υπέρ. Απορρίπτεται. 8 υπέρ. Απορρίπτεται. 9 υπέρ. Απορρίπτεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ. Απορρίπτεται. 11 υπέρ. Συγγνώμη. 11 υπέρ. Απορρίπτεται. 12 υπέρ. Απορρίπτεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Εγκρίνεται. 13 υπέρ. Απορρίπτεται. 14 υπέρ. Α, συγγνώμη λέει ο πρόεδρος. 20 υπέρ. Απορρίπτεται. 21 υπέρ. Εγκρίνεται. Συγγνώμη, 21 ας γίνει έλεγχος ηλεκτρονικός για την 21 ηλεκτρονική ψηφοφορία που ξεκινάει. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Το αποτέλεσμα είναι 23 με 23. Ίδια ισορροπία, ίδιος αριθμός ψήφων. Απορρίπτεται. Μόλις. Πάμε στην τροπολογία 22 υπέρ. Απορρίπτεται. 23 υπέρ. Απορρίπτεται. 24 υπέρ απορρίπτεται 25 υπέρ απορρίπτεται 26 και 27 υπέρ απορρίπτονται 28 υπέρ εγκρίνεται 29 υπέρ εγκρίνεται 30 υπέρ απορρίπτεται 31 υπέρ εγκρίνεται 32 υπέρ εγκρίνεται 33 υπέρ απορρίπτεται 34 υπέρ απορρίπτεται 35 υπέρ απορρίπτεται 6 υπέρ. Απορρίπτεται. 37 υπέρ. Απορρίπτεται. 38 υπέρ. Απορρίπτεται. 39 υπέρ. Εγκρίνεται. 40 υπέρ. Εγκρίνεται. 41 υπέρ. Απορρίπτεται. 1 υπέρ. Απορρίπτεται. 2 υπέρ. Απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε την γνωμοδότηση ίντε. Ψηφίζουμε την 1, 2, 3 μαζί υπέρ απορρίπτεται. Είναι τα 4 υπέρ, εγκρίνεται. Είναι τα 5, εγκρίνεται. Είναι τα 6 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, απορρίπτεται. Είναι τα 7 υπέρ, απορρίπτεται. Είναι τα 8 υπέρ, εγκρίνεται. Είναι τα 9 υπέρ, εγκρίνεται. Είναι τα 10 και 11 υπέρ, απορρίπτονται. Είναι τα 12 υπέρ, εγκρίνεται. Είναι τα 13 υπέρ. Απορρίπτεται. Είναι τα 14 με προφορική υπέρ. Εγκρίνεται, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε έκον. 1, 2 και 3 υπέρ. Απορρίπτονται. Έκον 4 υπέρ. Με προφορική εγκρίνεται. Έκον 5 υπέρ. Εγκρίνεται. Έκον 6 υπέρ εγκρίνεται. Έκον 7 υπέρ, εγκρίνεται. Έκον 8 υπέρ, εγκρίνεται. Έκον 9 υπέρ, απορρίπτεται. Έκον 10 υπέρ, εγκρίνεται. Έκον 11 υπέρ, εγκρίνεται. Έκον 12, 13 και 14 υπέρ, απορρίπτονται. Τελική λήξη και ψηφορία για το σχέδιο εκθέσεω που τροποποιήθηκε. Ξεκινάμε τη ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Τέλο ψηφοφορία. Και το αποτέλεσμα είναι 43 ψήφοι υπέρ, μία ψήφος κατά, μία αποχή. Συγχαρητήρια λοιπόν στον κύριο Μιλανμόν. Λαμπρό είναι το μέλλον μας στις διατηλετικές σχέσεις, χάρη στη δική σας έκθεση, κύριε Μον. Και περνούμε στο επόμενο σημείο, την, το σχέδιο έκθεσης και παρακαλώ θερμά όσους δεν πρόκειται να παραμείνουν στην αίθουσα για τη συζήτηση, να την εγκαταλείψουν ε, χωρίς πολύ θόρυβο, προκειμένου να περάσουμε στο σημείο 13 με θέμα την εδραίωση της σταθερότητας και της ευημερία στα Δυτικά Βαλκάνια. Η συγκεκριά μας είναι η κυρία Άννα Δευτό. Στην οποία και δίνω το λόγο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 Ευχαριστώ θερμά τους ευγενείς συναδέλφους που παρέμειναν στην αίθουσα για να παρακολουθήσουν τη συζήτηση. Θα παρακαλούσα τους ε, ενθουσιώδεις Ισπανούς εισαγωγή αποσιοποιητικά. Το λόγο έχει η Μπρισάντζιτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Mm har valt att i den här rapporten eh, vara ganska övergripande. Eh, det vill säga... Στην έκθεση αυτή Αναφέρομαι σε διάφορες άλλες εκθέσεις. Υπάρχει μια ολόκληρη σειρά άλλων εκθέσεων που πραγματεύονται το θέμα αυτό. Άρα διαμορφώνω οριζόντια, αν θέλετε, το θέμα αυτό, δεν αποφύγουμε και τις ε, επικαλύψεις. Ε, επικεντρώνουμε στα θέματα εκείνα τα οποία είναι κοινά για τις πιο πολλές χώρες των Ανατολικών Βαλκανίων. Και στη συνέχεια εστιάστηκα στα όσα θα έπρεπε να συμβούν προκειμένου να καταστεί δυνατή η προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έγινε μια πρώτη συζήτηση για την έκθεση αυτή στο Στρασβούργο και έλαβα πολύ θετικέ παρατηρήσεις και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα θετικά αυτά σχόλια και την καλή συνεργασία στο Στρασβούργο. Έλαβα πολλές ενδιαφέρουσες προτάσεις και άλλωστε ζήτησα να υποβάλλετε και τροπολογίες, τις περισσότερες εκ των οποίων μπορώ να υποστηρίξω. Νομίζω ότι τελικά θα καταφέρουμε να πετύχουμε πολύ καλούς συμβιβασμούς. Αρχικά σκοπός ήταν να υπάρξει προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών μόνο μία ημέρα. Ωστόσο, θεώρησα ότι ήταν πάρα πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα, γι' αυτό και προβλέφθηκε τελικά μία εβδομάδα. Αν θέλετε να υποβάλλετε τροπολογίε, έχετε ακόμα καιρό και ίσως θα μπορούσε να μας πει και η γραμματεία ποια θα είναι ακριβώ η προθεσμία. Εν πάση περιπτώσει θα είναι παραπάνω από μία ημέρα. Και αναφορικά με την παράγραφο 2 και 3 σίγουρα θα υπάρξουν συζητήσεις, Άλλωστε αυτά ήταν και τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν και την προηγούμενη φορά στην, ε, στο Στρασβούργο. Πρόκειται για τις παραγράφους που αναφέρονται στη συνθήκη της Λισαβόνας. Αρκετές χώρες έχουν και τηρούν επιφυλακτική στάση αναφορικά με περαιτέρω διεύρυνση. Θα ήθελα λοιπόν να διατηρηθεί αυτή η πρόταση ακριβώς για να γίνει η συζήτηση αυτή. Η έκθεση αυτή δεν περιλαμβάνει νέα στοιχεία, δεν περιλαμβάνει στοιχεία τα οποία δεν έχει αναφέρει άλλωστε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα όσα έγραψα έχουν ήδη αναφερθεί, αλλά κανένας ευρωπαϊκός θεσμός δεν το έχει θέσει έτσι σε χαρτί. Αυτό μπορεί να αποτελέσει αμφιλεγόμενο θέμα, το αντιλαμβάνομαι αυτό και γι' αυτό και είμαι διατεθειμένη να αναζητήσω συμβιβαστική λύση, αλλά θα ήθελα καταρχάς να το συζητήσουμε στην Επιτροπή και θα χαρώ να λάβω και τροπολογίες στη συνέχεια. Να τονίσω ιδιαίτερως κάποιες ε, δύο παραγράφους, τη 18 και τη 19 γιατί διαρκώς αναφέρουμε το πόσο σημαντική είναι η συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο προκειμένου να μην μένουν ατιμόρυτα τα διεθνή εγκλήματα. Και αναφέρεται κάτι το οποίο περιλαμβάνεται στο νόμο πολλών χωρών σχετικά με την έκδοση εγκληματιών σε δικαστήρια άλλων χωρών. Αυτή η απαγόρευση που περιλαμβάνεται συνεπάγεται μεγάλα προβλήματα αναφορικά με την εκδίκαση δηλαδή εγκληματιών πολέμου που έχουν διαπράξει διεθνή εγκλήματα από διεθνή δικαστήρια. Θεωρώ ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουν να υφίστανται αυτές οι απαγορεύσεις εθνικά, στην εθνική νομοθεσία. Αυτό και εκφράζω ουσιαστικά και στις παραγράφους αυτές. Υπάρχουν Υπάρχουν πολλά επιχειρήματα για την καταδίκη της απαγόρευσης αυτής και θα πρέπει με σαφήνεια να εκφράσουμε την άποψή μας αυτή ότι δεν είναι δυνατόν τα κράτη στα Βαλκάνια να διατηρούν τέτοιες νομοθεσίες οι οποίες δυσκολεύουν το έργο των διεθνών δικαστηρίων. Συνομίλησα και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με κάποια μέλη του Συμβουλίου δεν μπορεί να τεθεί τέτοια απέτηση πριν από ενδεχόμενη διεύρυνση. Ωστόσο, πρέπει να πω ότι δεν έχει γίνει ποτέ και διεύρυνση με χώρες που έχουν, στις οποίες έχει υπάρξει τέτοιος πόλεμος. Άρα τίθεται πλέον το θέμα και υπάρχουν, συντρέχουν οι λόγοι για να τεθεί τέτοιος όρος. Αυτό το θέμα λοιπόν της απαγόρευσης είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι δυνατόν να γίνει περαιτέρω διεύρυνση προτού εκδικαστούν οι εγκληματίες πολέμου. Αυτά λοιπόν και ανυπομονώ να ακούσω και τις συζητήσεις ε, και τις τροπολογίες σας. Αν ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Πριπέτης. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Ιμπρισάτζιτς για την έκθεσή της με θέμα την εδραίωση της δημοκρατίας, της σταθερότητας και της ευημερίας στα Βαλκάνια. Νομίζω ότι η ραχοκοκαλιά της έκθεσης αυτής ε, δεν μπορεί παρά να μας βρίσκει σύμφωνος. Δηλαδή, η διέξοδος ε, των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, δηλαδή η Κροατία πρώην δημοκρατία, δημοκρατία της Μακεδονία, Μακεδονίας, Φιρόμ, Σερβία, Αλβανία, δεν μπορούν παρά να έχουν μια ευρωπαϊκή προοπτική και μια διέξοδο, διέξοδο του στην ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης θα πρέπει να προσδιορίσουμε με σαφήνεια την περιφερειακή προοπτική αυτών των χωρών και να δώσουμε και τη δέουσα προβολή σε αυτή την προσέγγιση. Συμφωνώ επίσης με την ανάγκη να ξεπεράσουμε τις διμερείς συγκρούσεις, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της ενταξιακής διαδικασίας αυτών των χωρών. Χαίρομαι για την πρόταση επενδυτικού πλαισίου για τα Δυτικά Βαλκάνια και έχω κάποιες παρατηρήσεις ε, για το τι συνέχεια θα πρέπει να δοθεί στην έκθεση αυτή ανακύπτει καταρχήν το θέμα του ίδιου του μέλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί με τον ισχύοντα μηχανισμό, αν διευρυνθούμε σε 30 και παραπάνω χώρες, οι ισχύωσες διαδικασίες δεν είναι κατάλληλες. Δεν μπορούμε λοιπόν να ορίσουμε ένα πλαίσιο αν δεν εξασφαλίσουμε ένα θεσμικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που την καθιστά λειτουργική, ε, με αποτελεσματικές πολιτικές αλλά και με δράση, με ικανότητα απόφασης και δράσης. Επίσης, η κοινωνία γέννη και η κοινή γνώμη στις χώρες μας δεν ε, βλέπουν πάντα με καλό μάτι ε, τη διεύρυνση. Δεν θεωρούν ότι κάθε διεύρυνση είναι και μια ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αναδειχθεί σε παγκόσμιο εταίρο και να αναλάβει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο. Βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις ότι πολύ συχνά η διεύρυνση ε, θεωρήθηκε από, πολλές, ε, από πολλούς λαούς ως ε, μία ορμή προς τα εμπρός χωρίς να ληφθεί υπόψη όντως η γεωγραφική κατάσταση. Έτσι τη βίωσαν πολλοί πολίτες στη διεύρυνση. Δεν μπορούμε επίσης να προσδιορίσουμε μια διαδικασία χωρίς να την πρικοδοτήσουμε με δημοσιονομικά μέσα. Είναι σαν να ε, προσπαθούμε να επιδιορθώσουμε ένα σπίτι και να το μεγαλώσουμε χωρίς να βάζουμε το χέρι στην τσέπη για να χρηματοδοτήσουμε αυτές τις ε, επισκευές και τις διαβρύσεις. Θα πρέπει λοιπόν στο μέλλον ο προϋπολογισμός μας να είναι πιο ε, πλούσιος, όχι μόνο για να εφαρμόσουμε λειτουργικά τις ε, πολιτικές ένωσης, αλλά και να δώσουμε σάρκα και οστά στην προσδοκία, την εύλογη προσδοκία των ε, χωρών των Δυτικών Βαλκανίων για ένταξη μια μέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα παιδιτικό πλαίσιο για τα Δυτικά Βαλκάνια που θα συντονίζει όλα αυτά τα εγχειρήματα και θα πρέπει να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας και να πρικοδοτήσουμε τον προπολογισμό μας, με, τον προϋπολογισμό μας με μέσα αντάξια των ε, προσδοκιών μας. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Καζάκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ και εγώ απόλυτα με τον προλαλήσαντα. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγητριά μας για την άρτια έκθεσή της και να πω ότι κατά τη γνώμη μου τα Δυτικά Βαλκάνια είναι μια πολύ ευάλωτη περιοχή και εκεί τα γεωπολιτικά και στρατηγικά συμφέροντα πολλές φορές είναι συγκρόμενα, αποκλίνονται. Εξού και ο ευπαθής χαρακτήρας αυτής της περιοχής σε ό,τι αφορά την σταθερότητά της. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύω ότι θα πρέπει να προσέξει όλο και περισσότερο το θέμα της συνδρομής προς τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, ώστε να μπορέσουν οι χώρες περιφέρειας αυτής να εξασφαλίσουν τη σταθερότητά τους και να εστερνιστούν τις ευρωπαϊκές αξίες. Γι' αυτό και πιστεύω ότι και το χρηματοοικονομικό και το δημοσιονομικό πλαίσιο υποστήριξη προς χώρες αυτές θα πρέπει να περιστρέφεται γύρω από τρεις κύριους στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι η παροχή τεχνικής συνδρομής στοχοθετημένης και εστιασμένης κυρίως στον εξυγχρονισμό των υποδομών. Γιατί η βελτίωση των υποδομών είναι εκ των όνων κάνευ προϋπόθεση όχι μόνο για τις μελλοντικές επενδύσεις, αλλά και για την οικονομική σταθερότητα των χωρών. Δεύτερον, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε και την κοινωνία των πολιτών στις χώρες αυτές, προκειμένου να απαλληθούν τα αρνητικά στερεότυπα που είναι χαραγμένα στη μνήμη των πολιτών των λαών αυτών. Αυτό είναι απαραίτητο αν θέλουμε πραγματικά να θεραιώσουμε τη σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια και να εξαλείψουμε τους φόβους αναζωπήρωσης των παλιών συγκρούσεων που δίχασαν την περιοχή. Επίσης θα πρέπει να προσπαθήσουμε για τη διαθέτηση των κρεμόσων πολιτικών και νομικών συγκρούσεων. Και πιστεύω ότι η υποστήριξη αυτή για την διαθέτηση των συγκρούσεων με αποδεκτή από όλους λύση είναι πολύ σημαντική προϋπόθεση για να μπορέσουν οι χώρες αυτές να προχωρήσουν στις ε, προενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστούμε κύριε Καζάκ. Ο κύριος Σταμπάιτζη. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια, την κυρία Ιμπρασίτς, διότι είναι πολύ ισορροπημένη η έκθεση. και είναι σημαντικότατη και είναι πάρα πολύ επίκαιρη. Παρακαλώ, προσέξτε το εξή. Η γενική γραμμή είναι πολύ καλή της εκθέσεως. Ίσως χρειάζεται κάποια μικρορύθμιση το κείμενο να διορθώσουμε κάποια προβληματάκια. Ποιες είναι οι συνέπειες της χρηματοπιστωτικής κρίσεως και οικονομικής κρίσεως, της παγκοσμίου κρίσεως στην περιοχή αυτή. διότι πριν συνταχθεί αυτή η έκθεση η χρηματοπιστωτική κρίση δεν ήταν τόσο μεγάλη όσο τώρα. Ίσως αυτές οι χώρες είναι πολύ πιο ευάλωτες από άλλες χώρες της Ευρώπης. Ίσως γι' αυτό θα έπρεπε να επιστήσουμε την προσοχή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως επ' αυτού. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, ο ευάλωτος χαρακτήρας της περιοχής από την ενεργειακή άποψη. Θα θυμόσαστε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι κατά τη διάρκεια της συγκρούσεως μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, τι έγινε. Διεκόπη η παροχή του φυσικού αερίου, η Σερβία και άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων βρέθηκαν σε αρκετά δραματική και τραγική κατάσταση. Και η χώρα μου, παραδείγματος χάρη, η Ουγγαρία, βοήθησε τη Σερβία για να λύσει τα σοβαρότατα προβλήματά της. Τρίτον, νομίζω ότι θα έπρεπε να τονίσουμε την κύρωση της Συμφωνίας Σταθερότητας και Σύνδεσης, την κύρωση και υλοποίησή της. Τελευταίο σχόλιο. Δεν φταίει κυρία Μπισάτζιτς. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να είναι σύντομη έκθεση. Όμως βλέπετε το περιπλοκότερο θέμα είναι η σχέση μεταξύ των εθνοτήτων στην περιοχή. Και εντός των κρατών και μεταξύ των κρατών οι σχέσεις. Όπως είναι το αλβανικό πρόβλημα. Το θέμα της Μεγάλης Αλβανίας. Υπάρχουν πολλά προβλήματα και για το μελλοντικό κοινοβούλιο. Πιστεύω ότι θα χρειαστούν και άλλες λεπτομερέστερες εκθέσεις επί του θέματος. Διότι θα απαιτούσε ξεχωριστή έκθεση αυτό το πρόβλημα. Αυτό το θέμα είναι τόσο οξύ, τόσο περίπλοκο και τόσο δύσκολο, τόσο δυσεπίλητο. Όχι μόνο Βοσνία, Ζεγοβίνη, ε, Κωσυφοπαίδιο, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Τη συγχαίρω λοιπόν την εισηγήτρια και από την πλευρά μου θα υποστηρίξω την έκθεσή της διότι είναι πολύ καλή πολύ καλή δουλειά που έκανε σας ευχαριστώ πολύ Υπάρχουν συνάδελφοι που θέλουν να πάρουν το λόγο με θέμα αυτή την έξοχη έκθεση. Θα ζητήσω από την κυρία Μπρεσάτζιτς να ολοκληρώσει τη συζήτηση. Θέλετε να πείτε κάτι. Ο κύριος Ναζάρ θέλει να πει κάτι. Θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη αφορά τις αποστολές που αναφέρονται στην έκθεση. Αναφέρεται ότι στόχος της αποστολής πρέπει να επιτευχθεί ο στόχος, να επιτευχθεί πλήρως. Εκεί θα πρέπει να αναφέρουμε και ένα χρονικό πλαίσιο. Όχι πολύ συγκεκριμένο, αλλά κάποιο χρονοδιάγραμμα. Και αναφέρω εδώ πιο συγκεκριμένα το πρόβλημα του κοσυφαπεδίου για την απελευθέρωση από την ανάγκη προξενικής θεώρησης. Πέραν του ότι θα έπρεπε να δικός μας στόχος, θα έπρεπε να συστήσουμε στα κράτη-μέλη να βοηθήσουν τις πρεσβείες τους να διευκολύνουν τη διαδικασία χορηγήσεως θεωρήσεων. Διότι υπάρχουν πολλές αιτήσει σε όλες αυτές τις χώρες και ακόμα και ένα κανονικό αίτημα δεν μπορεί να διεκπαιρεωθεί λόγω προβλημάτων, λόγω έλλειψης οσοπικού. Και ένα άλλο σχόλιο, ήταν αναφέρθηκε η Αλβανία. Η παρούσα αλβανική κυβέρνηση έχει πετύχει πολλά, την τελευταία διετία τουλάχιστον, κάτι που αναγνωρίστηκε, διότι πρόκειται να συσταθεί, να πρόσκληση να προσχωρήσουν στο ΝΑΤΟ. Αυτά ήθελα να πω. Και τώρα στο τέλος, εφόσον είμαι τελευταίος, να συγχαρώ την εισηγήτρια για την έκθεσή της. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχει άλλος συνάδελφος που θέλει να μιλήσει. Η κυρία Ιμπρισάτζης. Α, συγγνώμη. Άννα, Συγγνώμη, να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον κύριο Σερβάντες. Θέλετε να πείτε κάτι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχουμε ελάχιστα να πούμε. Η έκθεση πιστεύουμε ότι είναι πολύ καλογραμμένη, άριστη διατύπωση και όπως ανέφερε και η συγγήτρια, με, από πολιτική προσέγγιση αναλύει το θέμα. και έρχεται και έγκαιρα και έκθεση. Θα είμαστε σε επαφή με την εισηγήτρια, θα προσπαθήσουμε να τη βοηθήσουμε να διατυπώσει την έκθεση με τον καλύτερο τρόπο, ούτω ώστε ε, να βοηθήσουμε στην ένταξη και την ολοκλήρωση αυτού του τμήματος της Ευρώπης. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Άννα Εμπρεσάτζιτς, η εισηγήτρια, έχει το λόγο. Jag kommer naturligtvis inte kunna hinna gå med genom precis varenda kommentar som jag har fått. Jag skulle... Φυσικά δεν μπορώ να απαντήσω σε κάθε ένα σχόλιο που ακούσαμε. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για όλες τις παρατηρήσεις σας. Γιατί πραγματικά ήταν πολύ ωφέλιμες. Ο κύριος Ταμπάτζη ανέφερε ότι ίσως να λείπουν κάποια στοιχεία από την έκθεση ακόμη. Προσπάθησα να συμπεριλάβω όσο πιο πολλά ε, σημαντικά στοιχεία μπορούσα, αλλά έχετε δίκιο έπρεπε να παραμείνει κάπως συνοπτική η έκθεση. Η έκθεση δεν μπόρεσα να επεκταθώ σε όλα τα θέματα. Αλλά θα υποβληθούν και τροπολογίες και σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, γιατί αποτελεί ένα από τα θέματα τα οποία με απασχολούν ιδιαίτερα και το θέμα των μη Γιατί ακούσαμε το θέμα, το πρόβλημα των εθνικών συγκρούσεων, εθνοτικών συγκρούσεων. Αυτό αποτελεί σίγουρα ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην έκθεση. Δεν είναι δυνατόν να μην συμπεριληφθεί σε μια τέτοια έκθεση το ζήτημα αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον πρώτο ομιλητή που είπε ότι η κοινή γνώμη στις χώρες μας δεν ε, συμφωνεί σε πολλές περιπτώσεις ε, με τις προοπτικές διεύρυνσης. Συμφωνώ, συμφωνώ και ακριβώς για αυτό το λόγο κατήρτισα την έκθεση αυτή έτσι. Όταν η κοινή γνώμη δεν καταλαβαίνει ποιες είναι όλες οι ωφέλειες, ε, ποιες είναι οι άμεσες συνέπειες της διεύρυνσης και τι θα σημαίνει αυτό για παράδειγμα αν δεν υπάρχει διεύρυνση για παράδειγμα τι θα σημαίνει αυτό για την ασφάλεια σε ευάλωτες περιοχές όταν λοιπόν ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει αυτό είναι καθήκον μας εμείς ε, ως πολιτική να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση και να εξηγήσουμε τα στοιχεία αυτά στο κοινό. Εμείς ως πολιτικοί πρέπει να κάνουμε τις συζητήσεις αυτές και με τον τρόπο αυτό νομίζω ότι δεν δίνουμε και τη σωστή προοπτική. Άρα νομίζω ότι συμπεριλαμβάνεται ήδη ε, παρκώς στην έκθεση. Αν θέλετε να το τονίσουμε το στοιχείο αυτό, ε, θα χαρώ να λάβω τις τροπολογίες σας. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, θα τις ε, υποστηρίξω. Τώρα, σε ό,τι αφορά το τομέα της χρηματοδότησης, θα πρέπει να υπάρξει και διεύρυνση της χρηματοδότησης. Συμφωνώ, δεν αφιέρωσα τόσο μεγάλο κομμάτι της έκθεσης ε, στη χρηματοδότηση γιατί το θεωρώ πολιτικό εργαλείο. Για μένα το θέμα ήταν το τι θέλουμε να πετύχουμε στην Ευρώπη. Και φυσικά και θα πρέπει να υπάρχουν τα ανάλογα κονδύλια, αυτό εννοείται. Κάποιοι συνάδελφοι στην Επιτροπή Προϋπολογισμών έχουν την εντύπωση ότι ίσως αυτό να μην ισχύει, ίσως να έχουν διαφορετική άποψη ίσως να θεωρούν ότι ήδη χρηματοδοτούνται πάρα πολλά, αλλά αν θέλουμε να δηλώσουμε πολιτικώς πώς τι θέλουμε να πετύχουμε στην Ευρώπη, θα πρέπει να βρούμε και τον τρόπο να το χρηματοδοτήσουμε. Αυτό που έχουμε θέσει ως πολιτική προτεραιότητα για τον κύριο Κάζακ. Ναι, όντως. Τα Δυτικά Βαλκάνια αποτελούν μια πολύ εύθραυστη περιοχή, μια ευάλωτη περιοχή. Είναι πάρα πολύ σημαντική όμως η περιοχή αυτή για την ευρωπαϊκή σταθερότητα παρακολούθησα πολύ στενά τις χώρες αυτές κάτι την πενταετή θητεία μου και όποτε έχουμε δώσει σαφή ευρωπαϊκή προεπτική στις χώρες αυτές, αυτό έχει οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Όποτε αποτυγχάνουμε εμείς, ακολουθούν εθνικιστικές τάσεις, εθνικιστικές επιλογές, οι οποίες ασφαλώς δεν είναι θετικές για το Μαυροβούνιο την ε, Μακεδονία, λέει ομιλήτρια, που θα διοργανώσει εκλογές σύντομα στην Κροατία, εκλογές το 2010 στη Σερβία και επιμένω, θα πρέπει να δώσουμε μια σαφή ευρωπαϊκή προοπτική. Αν θέλουμε οι χώρες να προσεγγίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση με τις ε, σχετικές ε, μεταρρυθμίσεις. Δεν θα ήθελα καν να σκεφτώ ποια θα ήταν η εναλλακτική λύση, γιατί θεωρώ ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση για τα Βαλκάνια. Και τα να αναφέρθηκα στα σχόλιά σα. Να επαναλάβω ότι αν έχετε πιο συγκεκριμένες προτάσεις για τα δικαιώματα των μειονοτήτων, αν θέλετε να υποβάλλετε συγκεκριμένες τροπολογίες, θα χαρώ να τις συμπεριλάβω, κυρία Νάσαρη, για τις αποστολές στην ε, περιοχή αυτή. Αυτό που έχω μάθει είναι ότι τα πράγματα είναι δύσκολα για τη Βοσνία, για παράδειγμα, όπου έχουμε και στρατηγικές και πολιτικές αποστολές. Αυτά δεν μπορούμε να τα ερθετήσουμε χρονικά, γιατί οι περιοχές αυτά, αυτές τροποποιούνται, αλλάζουν συνεχώς και σημαίνουν διάφορα αναπάντεχα περιστατικά. Και όταν, για παράδειγμα, ο ύπατος εκπρόσωπος στο Σαράγεβο αποκλείστηκε. Δεν ε, φανταζόμασταν τότε ότι η λύση για το Κόσοβο, για το Κωσυφοπέδιο, θα ακολουθούσε δύο χρόνια αργότερα. Και αναγκαστήκαμε να παρατείνουμε την ε, εντολή του ύπο του εκπρόσωπου στο Κωσυφοπέδιο. Αυτό δεν μπορούμε να το φανταστούμε και να το προβλέψουμε εκ των προτέρων. Αν, το είχαμε, παρατη... αν ε, προβλέψει μία συγκεκριμένη περίοδο θετίας. Δεν θα μπορούσε να έχει ακολουθήσει αυτή η εξέλιξη των περιστάσεων. Θα πρέπει λοιπόν διαρκώς να κάνουμε αξιολόγηση προκειμένου να παραμένει σταθερή η κατάσταση γιατί δεν θέλουμε φυσικά να φύγουμε από την περιοχή αυτή πολύ νωρίς. Επαναλαμβάνω ότι έζησα από κοντά τον πόλεμο και τα πράγματα είναι πολύ πιο ευάλωτα και ευαίσθητα από ό,τι φαντάζεστε. Άρα δεν ε, συστήνω να προτείνουμε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Να έχουμε μια φιλοδοξία. Μια φιλοδοξία με συγκεκριμένα benchmarking, προκειμένου να ξέρουμε ποια θα είναι το επόμενο βήμα μας. Σας ευχαριστώ και πάλι για όλες σας τις παρατηρήσεις και θα χαρώ να λάβω τροπολογίες. Ευχαριστούμε την εισηγητριά μας και όλους όσους έλαβαν μέρος στη συζήτηση. Η προθεσμία για την κατάσταση των τροπολογιών λήγει στις 3 Μαρτίου. Προχωράμε στο επόμενο θέμα της της διάταξης, το σημείο 14, την ενσωμάτωση της διάσταση του φύλου σε εξωτερικές σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση και στην αδρέωση τη ειρήνης και εθνική συγκρότηση. Πρόκειται για έκθεση του Αντιπροέδρου της ε, Επιτροπής μας, Λίμπο που για πολύ σοβαρούς λόγους ε, κολλείεται σήμερα. Αντικαθίσταται από την κυρία Ναπολετάνο, η οποία θα μας κάνει την παρουσίαση της έκθεσης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του συναδέλφου Ρούτσεκ που δεν μπόρεσε σήμερα να παρίσταται μαζί μας διότι είναι σε μια εξωτερική αποστολή και εγώ πρέπει να πω ειλικρινά σε εσά και στους συναδέλφους ότι χρησιμοποίησα τις σημειώσεις, τους, σημειώσεις του και τις πληροφορίες που μου έδωσε για να σας παρουσιάσω στη θέση του τις ε, γραμμές εκείνες που θα αποτελέσουν την έκθεση επί της οποίας θα πρέπει να αποφασίσει η Επιτροπή αυτή να την τροποποιήσει και να την εγκρίνει. Λοιπόν, οι διάφορες βάσεις από τις οποίες ξεκινά η έκθεση είναι ότι η διάσταση των φύλων στην εξωτερική πολιτική, της ότες των φύλων, ε, γίνεται όλο και πιο σημαντική διάσταση, κυρίως όσον αφορά την πρόληψη των συγκρούσεων, αλλά και την διαχείριση των τραγικών ε, περιστάσεων που επικρατούν μετά τις συγκρούσεις στη, στον ΟΗΕ τον ίδιο βασίστηκαν σε δύο θεμελιώδη ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Το πρώτο ψήφισμα του Οκτωβρίου του 2000 που αφορά ακριβώς το ρόλο των γυναικών στην ειρήνη και στην ασφάλεια και το δεύτερο ψήφισμα είναι πιο πρόσφατο του Ιουνίου του 2008 και αφορά τη σεξουαλική ε, βία ε, στις συγκρούσεις και στις καταστάσεις μετά τις συγκρούσεις. Δυστυχώς ε, ο, βιασμοί, ο βιασμός ήταν και είναι και θα είναι δυστυχώς ένα από τα μέσα του πολέμου, ένα μέσο ταπείνωσης του εχθρού. Τα σώματα λοιπόν των γυναικών θεωρούνται σαν αντικείμενα πάνω στα οποία ε, ξεσπάει μια βεντέτα και αυτό δημιουργεί φρικτές καταστάσεις για τη ζωή αυτών των ανθρώπων και τεράστιες επιπλοκές. Τούτων λεχθέντων είναι σημαντικό η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μια συνεκτική πολιτική η οποία θα έχει σαν στόχο να μπορεί να εφαρμόσει αυτούς τους προσανατολισμούς στο ΟΗΕ όσον αφορά την συμπερίληψη του θέματος ότες των φύλων σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας. Γι' αυτό η Επιτροπή μας, το Προεδρείο της Επιτροπής αποφάσισε να δώσει ζωή σε αυτή την πρώτη έκθεση που αφορά αυτή την πτυχή. Θα είναι η μόνη δυνατότητα για το Κοινοβούλιο να τοποθετηθεί επ' αυτής της διαστάσεως για την ανάπτυξη, τα πλαίσια της αναπτύξεως σχεδίων δράσεως. Το σχέδιο δράσεως που εξετάζουμε βασίζεται σε δύο πτυχές. Η πρώτη αφορά τις δεσμεύσεις, τα εξωτερικά καθήκοντα της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η άλλη πτυχή αφορά την εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το προσωπικό δηλαδή τους οργανισμούς και το πώς θα μπορεί να παρεμβαίνει σε τέτοιου είδους διακρίσεις στα πλαίσια της εξωτερικής πολιτικής. Αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό διότι δείχνει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συνοχή και συνέπεια σχετικά με τις δύο αυτές πτυχές. Και γι' αυτό χρειάζονται δείκτες όσον αφορά τις συγκεκριμένες πολιτικές που εφαρμόζονται, δείκτες και κίνητρα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την επίτευξη του στόχου να συμπεριληφθεί αυτή η διάσταση στις εξωτερικές σχέσεις. Θα πρέπει να υπάρχουν πόροι επαρκής οικονομικοί και πόροι που θα ταιριάζουν με τους ε, στόχους που θα πρέπει να πετύχουμε και θα πρέπει εμείς οι ίδιοι σε πιο συνολικό επίπεδο και σε πολύ ψηλό επίπεδο να εκφράζουμε αυτή τη δυνατότητα να υπάρχουν γυναίκες στο πιδάλιο του προσωπικού που ασχολείται ε, με τις αντιπροσωπείες, με το έργο των αντιπροσωπιών, με τις ειδικού αντιπροσώπους που εν γέννη αυτοί θεωρούνται στην, στο συλλογικό, στη συλλογική συνείδηση σαν θέσεις αντρικές. Η Αμερικανική κυβέρνηση πρόσφατα έλαβε παρόμοια μέτρα και βλέπουμε ότι οι γυναίκες δεν τα καταφέρνουν χειρότερα όσον αφορά την εξωτερική πολιτική και η κυρία Ολμπράιτ και η κυρία Κάρτερ ε, ελπίζω ότι θα εκπροσωπήσει πολύ καλά την πολιτική του Προέδρου και των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρέπει να κάνουμε και εμείς αντίστοιχα πράγματα. Και εμείς έχουμε κάνει μικρά πράγματα, έχουμε μια επίτροπο για την εξωτερική πολιτική, αλλά αυτό ακριβώς θα πρέπει να βοηθήσει την προετοιμασία του προσωπικού, ούτω ώστε να είναι όλο και πιο μεγάλη συμμετοχή των γυναικών στο προσωπικό των αντιπροσωπιών μας. Τέλος, ο εισηγητής θα ήθελε αυτό το έγγραφο, το πρώτο έγγραφο να αποτελέσει δικείμενο συζήτηση και να τροφοδοτήσει και τροπολογίε που υποβάλλουν οι συγητέ. Θα είναι πολύ ευτυχή ο συγητή να εξετάσει τι τροπολογίε των συναδέλφων και να τι συμπεριλάβει στην έκθεση. Τελευταία επισήμανση και πιο συγκεκριμένη είναι αυτή, η οποία αφορά και τα σχέδια δράσεων για να ευαισθητοποιηθούν τα κράτη-μέλη να λάβουν υπόψη αυτή τη διάσταση εξωτερική της πολιτική. Και αυτό είναι ένα σημείο που πονάει θα έλεγα, οδυνηρό, ακαθόδες, διότι κάποια κράτη-μέλη δεν φαίνεται να έχουν τέτοιες προθέσεις να εθετήσουν αυτή τη γραμμή παρόλο που αυτά που υπογραμμίζει ο εισηγητής δείχνουν ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη δεν έχουν εθετήσει με τέτοια προσέγγιση και τέτοια σχέδια δράσης. Η έκθεσή μας από τη στιγμή που θα εγκριθεί θα είναι χρήσιμη. Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κινητοποιήσει και να δώσει κίνητρα αν θέλετε στα κράτη-μέλη της Ενώσεως σχετικά με αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Ναπολετάνο. Οι στατιστικές μας δείχνουν, οι στατιστικές από την Επιτροπή Εξωτερικών, ότι 20% των μελών της Επιτροπής είναι γυναίκες. Ευελπιστούμε ότι θα αυξηθεί το ποσοστό αυτό στην επόμενη κοινοβουλευτική θητεία. η γραμματεία μας αντίθετα κυριαρχείται από γυναίκες. Θέλει κανείς το λόγο για την έκθεση Ρόουτσεκ με θέμα την εσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις εξωτερικές σχέσεις. Ουδής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μάλιστα, η προθεσμία για τις τροπολογίες λήγει στις 4 Μαρτίου. Τι άλλο να πούμε κύριε Ναπολετάνο. Ολοκληρώνεται η συζήτηση επί της εκθέσεως του σημείου 14. Έχω την Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας αναγγείλω μια διακοπή της συνεδρίας μέχρι τις 5.30. Περιμένουμε τον Γιάνν Κόχουτ, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, την Προεδρία στο Συμβούλιο για να μας ενημερώσει για την χθεσινή και προχθεσινή διάσκεψη υπουργών. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να έρθει λίγο νωρίτερα. Ας πούμε ραντεβού και πάλι στις 5 και 20 περιμένοντας τον Υφυπουργό της Τσεχικής